Λοιπόν, συνάδελφοι, αν συμφωνείτε, μπορούμε να συνεχίσουμε ε, με τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Ε, θα ήθελα να εγκρίνουμε πρώτα απ' όλα την ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, δεν έχω ανακοινώσεις να κάνω. Πάει και αυτό. Και Για να δούμε ε, πρώτα αν είναι εδώ ε, οι εισηγητές. Κυρία Μορέλ. Ο ε, κύριος Μάτο. Λοιπόν, ο κύριος Μάτο είναι εδώ παρόν. Ως εκ τούτου μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε και μόνο μία ώρα. Πρόκειται για ένα κοινό ε, σύστημα φόρου προστέμενης εξίσου όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφή επιβάρυνση σχετικά με τι παροχέ αγαθών και υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο. Ο εισηγητή είναι ο κύριο Μάτο. Παρακαλώ, κύριε Μάτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Η δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου, του κοινού ευρωπαϊκού χώρου, του ΦΠΑ, είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το σχέδιο δράσης και είναι απαραίτητο λοιπόν να βρούμε ένα σύστημα οριστικό για τον ΦΠΑ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το εμπόριο μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για να ξεπεράσουμε το σημερινό σύστημα το οποίο ήταν έτσι και αλλιώς μεταβατικό. Αν θυμόσαστε και σύμφωνα με αυτά που εγκρίναμε εδώ, αυτό το σύστημα οριστικό για τον φόρο προστιθέμενης αξίας βασίζεται ε, στην φορολόγηση στη χώρα ε, ε, αποστολής, ενώ το σημερινό σύστημα βασίζεται στην φορολόγηση στη χώρα από την οποία φεύγουν τα εμπορεύματα. Επειδή λοιπόν θα γίνει αυτή η μεγάλη αλλαγή, και μπορεί να χρειαστούμε πάρα πολύ χρόνο, αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάγκη παράλληλα να δούμε και μία ακόμα πρωτοβουλία που είναι αυτή τα επίγοντα μέτρα για να καταπολεμήσουμε την απάτη στα θέματα του ΦΥΠΙΑ και κυρίως ε, το γεγονός πως είναι μειωμένες οι εισπράξεις του ΦΥΠΙΑ. Αυτή η απάτη έφτασε τα 160 δις ευρώ, που είναι ανησυχητικό, και το διασυνοριακή αυτή απάτη είναι 50 δις ευρώ. Αυτό σε επίπεδο απώλειας φορολογικών εσόδων κατέτος. Και αυτές οι κινήσεις εμπορευμάτων διασυνοριακά είναι δύο ειδών. Καταρχήν το ένα είναι τροφοδοσία χωρίς ΦΠΑ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον αγοροπολισίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ΦΠΑ στη χώρα προς την οποία φεύγουν τα εμπορεύματα. Εδώ λοιπόν δίνεται η δυνατότητα να εγκριθεί για κάποια κράτη-μέλη να εφαρμόσουν προσωρινά ένα γενικευμένο μηχανισμό αντιστροφής ε, ε, του παθητικού ΦΠΑ, δηλαδή να μην το πληρώνει ο αγοραστής, αλλά ο προμηθευτής. Μεταβατικό σύστημα για συναλλαγές πάνω από τα 17.500 ευρώ. Στην πρόταση που είναι μια απλή πρόταση όπως έχετε δει και εσείς. Θέλουμε να διατηρήσουμε μια γραμμή παράλληλα, παράλληλα με αυτή του Συμβουλίου, δίνοντας όμως και μια σειρά ε, δικλειδών ασφαλείας που είναι απαραίτητες. Δηλαδή, θα χρησιμοποιούν το μέτρο αυτό μόνο τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν ε, απώλειες συλλογής ΦΠΑ υψηλότερο κατά 5% από το ευρωπαϊκό μέσο. Επίσης, πως θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα εγκρίνει τη χρήση αυτού του συστήματος και επειδή είναι μεταβατικό θα πρέπει να υπάρχει και ημερομηνία λήξη που θα είναι ο, Ιούνι, ο Ιούνιος του 2022 με ένα πειραματικό project που θα έλεγε επαναλαμβάνω το 2022. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε αυτές τις γραμμές μπορεί να λειτουργήσει, θα είναι ένα πιλωτικό σχέδιο, αλλά θα πρέπει να διατηρήσουμε ξεκάθαρο πως θέλουμε να εξασφαλίσουμε τα εξής δύο σημεία που είναι ουσιαστικά. Καταρχήν, η απάτη στο ΦΠΑ να μην μεταφερθεί απλώς από ένα κράτος μέλος σε κάποιο άλλο, δηλαδή να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο σημείο αυτό. Και δεύτερον, να μην παραλύσει με τον τρόπο αυτό η κοινή προσπάθεια που γίνεται και που θα πρέπει να συνεχίσει για να προχωρήσουμε προς ένα οριστικό σύστημα για το φόρο τη θέμενη αξία στην Ευρώπη. Αυτές είναι οι δύο βασικές αρχές, νομίζω των οποίων ε, όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ξέρω πως υπάρχει κάποια πολιτική ομάδα που δεν είναι υπέρ αυτών των θωμάτων, αλλά ξέρω πως θα συνεργαστούν μαζί μας, γιατί με τους σκιώδεις εισηγητές θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία και θα ξεκινήσουμε ήδη με ταχύ ρυθμό αν δεν αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν επιθυμεί κάποιος να λάβει το λόγο από τους σοσιαλιστές. Η κυρία Περέσο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να θυμόμαστε ότι ο φάκελος αυτός έχει μπλοκαριστεί εδώ και δύο χρόνια από ένα κράτος μέλος στο Συμβούλιο βάση της αρχής της ομοφωνίας, επειδή δεν έχουμε οριστικό καθεστώς ΦΠΑ, ο καθένας προσπαθεί να βρει μέσα, να βγει από την δυσκολία σχετικά με την απάτη. Το σύστημα αυτό του μηχανισμού παρουσιάζεται σαν ένα σύστημα ενδιαφέρον, πράγμα που εμείς δεν πιστεύουμε ως σοσιαλιστική και δημοκρατική ομάδα. Νομίζουμε ότι η καταπολέμηση της απάτης είναι να έχουμε ένα καθεστώς οριστικό. Στο Συμβούλιο, φάκελος αυτός, άλλοι φάκελοι ε, ΦΠΑ ε, παρεμποδίστηκαν για να έχουμε αυτόν τον μηχανισμό προς όφελος ενός κράτους μέλους. Καταλαβαίνουμε ότι ο συγητής ε, εμπνέεται από τη συμφωνία έτσι όπως συνάφθηκε στο Συμβούλιο, αλλά δεν βλέπω γιατί ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς πρέπει να υποστούμε αυτή την ομοιρία κατά κάποιο τρόπο στο, στο Συμβούλιο του Συμβουλίου και δεν νομίζω ότι εμείς έχουμε τάση να υποστηρίξουμε αυτό το μηχανισμό αυτοεκαθάρισης που δεν είναι κάτι το χρήσιμο για το μέλλον, παρόλο που η συμφωνία στο Συμβούλιο είναι μια συμφωνία προσωρινή, αλλά εφόσον δεν μπορώ να πω ποια θα είναι η θέση την οποία θα προτείνει ο εισηγητής στην ομάδα μας. Ευχαριστώ πολύ για το ECR Token. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να πω ότι χαιρετίζω το βήμα που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έννοια ότι πιστεύω ότι είναι σωστό ε, τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν ένα γενικευμένο μηχανισμό αντιστροφής επιβάρυνσης, να μπορούν να το πράξουν αν το επιθυμούν. Πρόκειται λοιπόν για ένα σημαντικό ελπιδοφόρο εργαλείο για την αντιμετώπιση του ΦΠΑ. Γνωρίζουμε ότι η διασυνοριακή αυτή απάτη έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει επιγόντως κάτι να γίνει. Ως εκ τούτου την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, την αντιμετωπίζω κάπως επιφυλακτικά που λέει ότι αυτός ο μηχανισμός ε, να εφαρμόζεται μόνο εφόσον η απάτη έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο, ένα επίπεδο το οποίο να κρίνεται ανησυχητικό. Κατά την άποψή μου, αυτό θα πρέπει να βρίσκεται στη διακριτική ευχαίρεια του κάθε κράτους μέλους. Το κράτος μέλος να κρίνει ε, κατά πόσον ε, ε, πρέπει να εφαρμόσει αυτό το γενικευμένο μηχανισμό. Και αν δηλαδή το κράτος πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να ελέγχει καλύτερα τα προβλήματα, τότε το, πρά το κράτος να μπορεί να το πράξει. Βεβαίως το θέμα είναι πώς αυτό το σύστημα θα είναι συμβατό με τα συστήματα άλλων κρατών μελών, αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι οποτεδήποτε εμφανίζονται προβλήματα θα μπορούσαμε να αναστείλουμε ε, αυτήν την ε, εφαρμογή. Αλλά ξέρετε κάτι, και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι εδώ για να αναστέλει πράγματα, αλλά για να καταθέτει προτάσεις για το πώς είναι δυνατόν να επιλύονται προβλήματα. Και υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, ε, όχι μόνο παρέκκληση από αυτό το μηχανισμό. Εγώ θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο μέχρι το 2022 είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, θα υπάρχει κόστος προσαρμογής, όχι όχι μόνο για το κράτος, αλλά και για τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει, όπως σας είπα, να υπάρχει παράταση και μετά το 2022. Αυτά είχα να σας πω και ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την έκθεσή του. Ξέχασα να το πω στην αρχή. Ευχαριστώ για την Άλντε Πίτερ Γέζεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω υποστήριξη για την προτινόμενη οδηγία που θα βοηθήσει ορισμένα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την φορολογική απάτη ε, με την ευθύνη αναφοράς ε, του, του ΦΠΑ και την ευθύνη του προμηθευτή. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες διότι δεν έχουμε χρόνο, απλώς θα περιοριστώ στο να πω ότι λόγω των ε, συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων ε, για το καθεστώς ε, ΦΠΑ, ίσως θα πρέπει να περιορίσουμε την εφαρμογή του γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης. Άκουσα τι είπε ο Λούκας, ότι ίσως θα πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο, δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον το Συμβούλιο πρότεινε να περιορίσουμε τον μηχανισμό ε, να τον, ως το 2022. Πρέπει ένα θέμα να το προσδιορίσουμε ως προς τη θέση του Κοινοβουλίου και εκεί συμφωνούμε με την πρόταση στο σχέδιο έκθεσης ότι η Κομισιόν θα λάβει την τελική απόφαση για το εάν ένα κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει τον μηχανισμό το Συμβούλιο εδώ και πάρα πολύ καιρό αγωνίζεται για το θέμα αυτό, έχει καταλήξει σε διάφορες συμφωνίες και θα πρέπει να είναι το Συμβούλιο που θα λάβει την τελική απόφαση βάσει πρότασης της Επιτροπής. Εγώ μάλλον υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση. Και τέλος πιστεύω ότι η θέση του Συμβουλίου περιλαμβάνει αρκετές διασφαλίσεις ρήτρες ασφαλείας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι ε, κάθε εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβράδυνσης δεν θα ε, θίξει ε, την ενιαία αγορά και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να, να είναι ευνοϊκό απέναντι στην θέση της Επιτροπής. Θα πρέπει η δική μας Επιτροπή να εργαστεί γρήγορα πάνω στο ε, φάκελο για να έχουμε μια θέση μέχρι το Δεκέμβριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ε, συμφωνούμε με την ανησυχία που υπάρχει ότι θα χάνονται εισοδήματα από τις ε, έσοδα μάλλον από τις απάτες ΦΠΑ και ότι θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις για να αντιμετωπιστεί η απάτη αυτή. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ένα οριστικό καθεστώς και γι' αυτό εμείς ε, στηρίζουμε αυτόν τον προσωρινό μηχανισμό της αντιστροφής της επιβάρυνσης κυρίως στους τομείς εκείνους όπου υπάρχουν βάσιμες υποψίες περί απάτης. Ε, τον γενικεμένο μηχανισμό. Μέχρι τώρα δεν τον έχουμε δεχτεί. Πρώτον, για οικονομικούς λόγους, διότι αυτός ο μηχανισμός αντιστροφή ε, δημιουργεί στρεβλώσεις ε, στα πλαίσια ενό γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφή επιβάρυνσης. Υπάρχει μια ολόκληρη οικονομική αλυσίδα. Μετακυλείται το βάρος στου καταναλωτέ. Η Κομισιόν έχει αναγνωρίσει ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν έχει την, το μηχανισμό αστυνόμευση του ισχύοντο συστήματο συστήματος του ΦΠΑ, όπου έχουμε πολλούς ε, μικρούς ε, και αυτοί φορολογούνται μέσα στην οικονομική αλυσίδα. Επιπλέον μπορεί να προκύψει άλλη μορφή απάτης ε, και θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό αντί να εξαλείψουμε γενικά την απάτη, η απάτη απλά να μετακυληθεί σε γειτονικέ χώρες ε, με τη μορφή χιονοστημάδας ε, και ε, κάποια κρατημέλη θα εφαρμόζουν το μηχανισμό της αντιστροφής, αλλά πάλι όχι. Θεωρούμε λοιπόν ότι ένα στοχευμένος μηχανισμός είναι χρήσιμος. Πιστεύουμε ότι η γενίκευση του συστήματος δεν θα λύσει το πρόβλημα, θα δημιουργήσει περισσότερους κινδύνους. Εμείς συμφωνούμε με την άποψη Επιτροπής που λέει ότι η καλύτερη επιλογή είναι ε, μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να επιβαρυνθούν επιχειρήσεις ε, και να παραμείνουν τα βασικά χαρακτηριστικά του ισχύοντος συστήματος FIPA. Αυτή την πρόταση θεωρούμε ότι δεν την εκρίνουν πολύ για καθαρά πολιτικούς λόγους. Δεν θέλουν δηλαδή να υπάρχει ένα αρμονισμένο καθεστώς FIPA στην κοινή αγορά. Συμφωνώ με αυτά που είπε η Περβά ότι δεν θα πρέπει να είμαστε όμοιροι ε, για αποφάσει που θα λάβει το Συμβούλιο για καθαρά πολιτικού λόγου. Έχουμε διαπιστώσει ότι η αρχή τη Ομοφωνία χρησιμοποιείται για να μπλοκαριστούν κάποιε αποφάσει ε, και κάποια κράτη έχουν δυνατότητα του βέτο. Ε, αυτό όμω είναι απαράδεκτο. Εμεί θα προτείνουμε τροπολογίε σε αυτή την πρόταση. Βέβαια, τελειώνετε σα παρακαλώ. Είχατε δύο λεπτά και έχετε ξεπεράσει. Ε, το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας. Ε, θέλω να σας πω ότι απλά εμείς θα συμμετέχουμε με καλό, θετική διάθεση στις ε, συζητήσεις. Η κυρία Ματίας, Α, δεν θέλετε το λόγο, ωραία. Η Μπάρμπερα Κάπαλ. Πρόεδρε, χαίρομαι για αυτή την πρόταση που κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θεωρώ ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα αν έχει κανείς κατά νου ε, το ύψος της απάτης και γι' αυτό ε, στηρίζω ανεπιφύλακτα το να εφαρμόζεται κάτω από ορισμένα κριτήρια ένας ε, μηχανισμός ε, αντιστροφής της ε, επιβάρυνσης. Γιατί πραγματικά μιλάμε για αυτό το φαινόμενο καρουσέλ, το οποίο φτάνει και μέχρι το 25%. Ο μηχανισμός αυτός βέβαια θα σημαίνει πολύ μεγάλη διοικητική επιβάρυνση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Τώρα, κατά πόσον θα πρέπει να εφαρμοστεί ο μηχανισμός αυτός μέχρι το 22% δεν ξέρω ξέρω. Επ' αυτού θα πρέπει να συζητήσουμε. Σε γενικές γραμμές ε, θεωρώ ότι ο κανισμός αυτός ε, που πρέπει να εφαρμοστεί θα αποφέρει μεγαλύτερα έσοδα στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό και γι' αυτό προσβλέπω σε μια ιδιαίτερα αγαστή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν ζητάει άλλο το λόγο, μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή. Ο κύριος Μάτος, ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ όσους πήραν το λόγο και να σας πω το εξής. Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία τα οποία συμμεριζόμαστε όλοι μας. Όλοι θέλουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι οριστικό. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις για το πόσο θα είναι η μεταβατική περίοδος, για παράδειγμα. Ε, και εκεί δεν μπορώ να συμφωνήσω με τα όσα είπε η κυρία Μπερέσου αλλά και κάποιοι ακόμα συνάδελφοι και θα σας εξηγήσω γιατί. Ναι, εμείς απορρίπτουμε το Συμβούλιο να μπορεί να μας βάλει βέτο ή να μας πιέσει, αλλά είναι προφανές πως εμείς δεν είμαστε μεν σε ομοιρία, αλλά θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο εξόδου από μια κατάσταση η οποία υπάρχει ε, και νομίζω ότι εδώ τα καταφέρνουμε. Βάζουμε κάποιους περιορισμούς, καταρχήν χρονικούς. Εσείς στηρίξατε το εξής. Ο κύριος Λούκε. Θα πρέπει να έχουμε αυτή την προθεσμία αλλά να μην δώσουμε υπερβολικά πολύ χρόνο, γιατί με τον τρόπο αυτό ίσως χάσουμε τη βούληση, την ευκαιρία ή και την δυνατότητα να δημιουργήσουμε αυτό το τουριστικό σύστημα. Οπότε, κάποια από τα θέματα τα οποία είναι στο τραπέζι, πρέπει να σας πω πως ουσιαστικά ξεπερνάμε τα προβλήματα με κάποιες από τις δικλείδες που προσφέρουμε μέσω του κειμένου. Οπότε πιστεύω Δεν έχουμε βέβαια την τελική λύση τώρα, αλλά Μέσω του συστήματος που προτείνουμε, πιστεύω ότι δίνουμε ένα μηχανισμό που θα μας επιτρέψει αυτή τη στιγμή να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και για το γεγονό ότι μπορεί να δημιουργήσουμε νέους, μεθόδου μεθόδους απάτης ε, ή να μεταφερθεί σε άλλα κράτη-μέλη απάτη με τις δικλείδες ασφαλεία που έχουμε εντάξει στο κείμενο, πιστεύω πώ θα το αποφύγουμε. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρχει αυτή η γενικότερη θετική προσέγγιση και χαίρομαι που οι χρονικές προθεσμίες θα μας οδηγήσουν στο να κλείσουμε το θέμα πριν τα τέλη της χρονιάς. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι ανοιχτό και σε οποιαδήποτε πρόταση, από οποιαδήποτε ομάδα, ακόμα και από αυτούς οι οποίοι δεν προτιμούν να δημιουργήσουμε αυτό το μηχανισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ το χρονοδιάγραμμα προθεσμία 5 Νοεμβρίου για τις τροπολογίες στις 5 το απόγευμα ε, εξέταση 26-27 Νοεμβρίου και μετά ψηφοφορία στην Econ. Θα πρέπει τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο, αλλά θα έρθει ε, βεβαίως ο εισηγητής διότι μιλάει στην Ολομέλεια θα έρθει τώρα σύντομα, γι' αυτό διακόπτουμε για λίγο περιμένοντας τον εισηγητή. Είναι ο ίδιος ο εισηγητής που λείπει. Θέλετε, κανείς, κάποιος από εσά να αντικαταστήσει τον κύριο Λούς. Βέβαια στο σημείο αυτό θα άρχιζε στις 8 και 20. Γι' αυτό υποθέτω ότι θα έρθει σε ένα λεπτό. Α, ήρθε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Um, λοιπόν, τώρα περάσαμε στο σημείο 6, κανόνες με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόλεψη, ανείχνευση, διερεύνηση, δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων. Ο εισηγητής είναι ο Σάντερ Λούς και είμαστε εδώ για να εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης του ε, για τη ΛΥΜΠΕ. Έχετε τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε με ε, συγχωρείτε πρέπει να μιλήσω στην Ολομέλεια. Θα προσπαθήσω να μην χρησιμοποιήσω τα τέσσερα λεπτά και να είμαι σύντομος. Είναι ένας φάκελος για την έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικές πληροφορίες. Αυτό είναι σημαντικό για τις ποινικέ έρευνες. Έχουμε το άρθρο 7.2 ε, και 2.10 είναι νομίζω τα άρθρα που βρίσκονται στον πυρήνα της πρότασης ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε αρμόδιες άρχες, ε, Europol κλπ. Και κάθε φορά που εξετάζουμε το θέμα αυτό, το θέμα που τίθεται θα έχουμε υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε αυτούς τους φορείς και αν έτσι είναι η περίπτωση θα έχουμε ωραίες μενες εξαιρέσεις ή θα είναι το αντίθετο, θα έχουν όλοι δικαίωμα ανταλλαγής πληροφοριών και αυτή η ανταλλαγή δεν θα είναι υποχρεωτική και ο καθένας θα μπορεί μόνος του να αποφασίσει. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μια διτή προσέγγιση, αλλά βεβαίως ε, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη των διαφόρων σκιωδών εισηγητών. Ε, είμαι ανοιχτό ως προς το θέμα αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία άρθρα, 7, 9 και 10. Άρθρο 7, το αίτημα, η αίτηση ε, στην ε, μονάδα οικονομικών πληροφοριών ε, ήθελε μια η Επιτροπή μια μαξιμαλιστική προσέγγιση χωρίς να λάβει υπόψη ε, την επιχειρησιακή ανεξαρτησία των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι ένα θέμα σημαντικό. Αυτή η λειτουργική ανεξαρτησία δεν ε, τονίστηκε μόνο στην οδηγία κατά του ξεπλήματος ε, βρώμικου χρήματος, γι' αυτό θα πρέπει να περιλάβουμε κάτι στην πρόταση αυτή, κυρίως όταν η ανταλλαγή ε, πληροφοριών θα μπορούσε να δείξει ποινικέ έρευνες ε, οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις μονάδες οικονομικών πληροφοριών και τα κράτη-μέλη και από την άποψη αυτή θα ήθελα να τονίσω ότι καταρχή υποστηρίζω την αρχική πρόταση της Επιτροπής ε, για την ενίσχυση αυτής ε, της ανταλλαγής ανάμεσα στις μονάδες χρησιμοποιώντας τα δίκτυα των μονάδων αλλά νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή είναι καλό να έχουμε κάποια διατύπωση για την κατάσταση, για τους όρους, για το πώς οι μονάδες θα χρησιμοποιήσουν αυτές ε, τις ε, πληροφορίες. Επίσης, η εμπιστοσύνη μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών ε, πληροφοριών για να ξέρουν για τι σκοπό θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες. Γι' αυτό πρότεινα μερικέ τροπολογίες σχετικά με την διατύπωση, ε, ανακολουθώντας ένα άρθρο της οδηγίας ε, κατά της ε, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ανάμεσα τώρα στις μονάδες και στην Europol, από την άποψη αυτή μπορώ να είμαι ε, σύντομος. Ε, δεν τροποποιήσαμε το άρθρο αυτό, διότι υποστηρίζουμε στενή συνεργασία ανάμεσα στις ομονάδες και την Europol. Η χώρα μου, το Βέλγιο, έχει πολύ καλή ε, συνεργασία με την Europol. Για όλα αυτά τα σημεία, βεβαίως, το θέμα που τίθεται είναι αν η συνεργασία θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Και θέλω να έχω τη σχόλιά σας ε, σε ε, τα θέματα αυτά. Δεν χρησιμοποίησα τα τέσσερα λεπτά, όπως βλέπετε, για την ομάδα του ΕΛΚ Μάρκους Βέρμπερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω εκ μέρους του κύριου Καντελάρη γιατί δεν μπορεί να παραστεί σήμερα. Θα συγχαρώ τον συνάδελφο και να σας πω πως πολλές φορές έχουμε επιμείνει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ταχεία και εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ε, αρμοδίων αρχών και στις ακρόασει για τα φορολογικά έχουμε πει πω υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των σχετικών μονάδων ε, των ε, οικονομικών desk και των αρμοδίων αρχών για θέματα φορολογικά, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να καταπολεμήσουμε και το ξέπλυμα και την τρομοκρατία και πολλές φορές ε, το να μην έχουμε αυτές τις πληροφορίες σημαίνει πως χάνουμε την ευκαιρία του να παρακολύσουμε κάποιου τέτοιου ε, ε, είδους εγκληματικές δράσεις και δημοκρατικές επιθέσεις και κάποιες έρευνες καταλήγουν σε αδιέξοδο γιατί ακριβώς δεν έλαβαν τα απόλυτα πλήρη στοιχεία στα πλαίσια των ερευνών τους. Οπότε, ο συνάδελφος που μου ανέθεσε να παρουσιάσω τις απόψεις τους, χαιρετίζει αυτές τις προσπάθειες έτσι ώστε να έχουμε όλοι ως αρμόδιες αρχές την πρόσβαση στα κεντρικά αρχεία αυτών των πληροφοριών, αλλά ο Τόμανς επίσης μιλάει για το θέμα ε, της σύστασης των σχετικών αρμοδίων μονάδων ε, στα κράτη-μέλη και το γεγονός πως αυτές θα πρέπει να διατηρήσουν την αυτονομία τους. Χρειάζεται λοιπόν να πετύχουμε μια ισορροπία μεταξύ αυτών των υπηρεσιών, των θεσμικών σωμάτων, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η καταστολή αυτών των εγκληματικών δράσεων. Οι τροπολογίες λοιπόν θα μιλήσει για τις δικαιοδοσίες οι οποίες ανταποκρίνονται στα αιτήματα για ενημέρωση έτσι ώστε να λαμβάνονται οι πληροφορίες με τρόπο που θα ευνοεί τις έρευνες εκτός από τις περιπτώσεις όπου θα είναι δυσανάλογες οι επιπτώσεις της αποκάλυψης σε φυσικό πρόσωπο ή ασχετές με το αντικείμενο για το οποίο έχουν ζητηθεί. Τέλος, ο επόπτης ε, για την προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησε για την ε, ανάγκη προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της ανταλλαγής ε, πληροφοριών μεταξύ των οικονομικών μονάδων, των δικαιοδοσιών και των αρμοδίων αρχών. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκ μέρου των σοσιαλδημοκρατών. Ε, ποιος άλλος, ποιος άλλος. Σκληρή ζωή και των συντονιστών ε, και των ε, πρόεδρων. Ο συνάδελφός μου και εκείνο ε, ζητά συγγνώμη γιατί δεν μπορεί να παρευρεθεί για λόγους τεχνικούς. Οι σοσιαλδημοκράτε χαιρετίζουν θερμά την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για βελτιωμένη πρόσβαση σε πληροφορίε σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρέ ποινικέ ε, πράξεις, ποινικά δικήματα. Το πλαίσιο, το νομικό που υπάρχει για να υπάρχει πρόσβαση σε οικονομικής φύσεως πληροφορίες ε, δεν είναι ικανοποιητικό για να αντιμετωπιστεί ε, το, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητε, μεταξύ άλλων και αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της, ε, ε των ε, για την υπόθεση των Panama Papers. Χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα παρακολουθεί και θέλει να εφαρμόσει και να υιοθετήσει νομοθετικές πράξεις. Ε, ο εισηγητής της ΕΚΟΝ προτείνει μια νέα διατύπωση για το πώς αυτή η νέα οδηγία θα προβλέπει τη συνεργασία ανάμεσα στις μονάδες οικονομικών ε, πληροφοριών ε, και σε άλλους ε, εμπλεκόμενους. Η μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις αρμοδιότητες αυτών των μονάδων και την, τα νομικά κριτήρια που ισχύουν προτείνουν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία, αυτό που προβλέπει και η πρόταση Επιτροπής. Όμως εμείς ανησυχούμε ε, για το ότι ο εισηγητής ε, σε αρκετές περιπτώσεις περιορίζει την αποτελεσματικότητα της οδηγίας προβλέποντας συγκεκριμένες διατάξεις. Αν θέλετε αυτό είναι ένα είδος ε, προσέγγισης που είχαμε προβλέψει στην Επιτροπή για τα Panama Papers, αλλά δεν θέλουμε να επαναληφθεί ε, σε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Ω εκ τούτου, οι σοσιαλδημοκράτες θα καταθέσουν τροπολογίε για να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία ανάμεσα στις οικονομικές αυτές μονάδες ε, και τις αρμόδιες ε, αρχές για να διευκολύνεται ε, η πρόσβαση. Ο Σκιώδης εισηγητής μας προσβλέπει σε επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή και με άλλες ομάδες για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, έτσι λοιπόν, τώρα πλέον δεν βλέπω να είναι παρόντες οι φιλελεύθεροι, η Ευαγγελή εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, σχέδιο γνωμοδότησης. Είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ε, την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οικονομικά εγκλήματα και διάφορα ποινικά αδικήματα. Σύμφωνο με την τον εισηγητή ε, να συμπεριλάβουμε εξαιρέσεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις μονάδες χρηματοοικονομικών ε, πληροφοριών και των αρχών, διότι ίσως μπορεί αυτό να έχει συνέπεια αρνητική όσον αφορά σε τρέχουσες έρευνες. Είναι σημαντικό να μην έχουμε πολύ αυστηρές υποχρεώσεις για τις μονάδες αυτές. Τελειώς αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό σε σχέση με το στόχο μας και ε, που θέλουμε να ενισχύσουμε την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος για να μην υπάρχει κακή χρήση οποιαδήποτε άρνηση σε αίτηση πληροφοριών πρέπει να αιτιολογείται Επίσης, σημερίζουμε την ανάγκη να προσθεθεί μια παράγραφος για να ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές να δίνουν ένα feedback, να απαντούν στις μονάδες αυτές σχετικά με την χρήση των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί και ως ε, προς το αποτέλεσμα της έρευνας και της δίωξης. Αυτό θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την συνεργασία ανάμεσα στις μονάδες αυτές και τις αρμόδιες αρχές. Νομίζω ότι κάτι λείπει. Κάτι λείπει από το σχέδιο γνωμοδότησης είναι ε, να έχουμε μία μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών που να είναι ευρωπαϊκή. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μία τέτοια μονάδα και ρόλος της θα ήταν να διευκολύνει τη συνεργασία και ακόμη και την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις μονάδες αυτές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, βεβαίως προσβλέπω στην ε, συνεργασία με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για να έχουμε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω την ΚΟΕ, εκπρόσωπο την ΚΟΕ και περνάμε στην διαδικασία Catch the Eye, ο εισηγητής όμως πρώτα. Πολύ σύντομα να πω ότι περιμένω με χαρά τις συζητήσεις που θα γίνουν και πιο συγκεκριμένα για τους πρασίνους ΕΛΚ και σοσιαλιστές. ΕΛΚ, νομίζω πως σας εμπνέει και η οδηγία κατά του ξεπλήματος που είναι καλό για μας και ενδιαφέρον. Οπότε με μεγάλη χαρά θα συνεχίσουμε και τη συζήτηση. Και για τις παρατηρήσεις της κυρίας Μπερές δεν σκοπεύουμε εμεί να αποδυναμώσουμε τη συζήτηση για την ανταλλαγή πληροφοριών, οπότε με χαρά θα δω με ποιο τρόπο θα ενισχύσουμε τις απόψεις ε, αμφότερων. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και για τους πράσινους να πω πως χαιρετίζουμε τα σχόλια για τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού θεσμού, μιας νέας υπηρεσίας. Αλλά βέβαια εδώ χρειάζονται κάποια ακόμα βήματα πριν φτάσει εκεί η συζήτηση. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στη συνάντηση των ε, σχεδόν εισηγητών. Μάλιστα. Το χρονοδιάγραμμα λέει 6 Νοεμβρίου για τις τροπολογίες της 5, συζήτηση τροπολογιών 26 και 27 Νοεμβρίου και ψηφοφορία σε εκείνη τη συνεδρίαση. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο. Είναι Θέσπιση προγράμματο για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικά των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβάνων των μικρομεσαίων και τι ευρωπαϊκέ στατιστικέ. Και έχουμε εδώ εισηγητή και πάλι τον κύριο Λούνε Σάντερ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα θέμα που συζητάμε ε, και έχει να κάνει με το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά που συγκεντρώνει κάποιες δράσεις που στο παρελθόν χρηματοδοτούνται από πέντε διαφορετικά προγράμματα με διαφορετικές γραμμές στον προπολογισμό και συμπεριλαμβάνει και κάποιες νέες πρωτοβουλίες για να λειτουργεί καλύτερα η εσωτερική αγορά. Αυτό είναι το πεδίο εφαρμογή και δεδομένου το ότι όλε αυτέ οι δράσει σχετίζονται με την ενιαία αγορά, είναι λογικό να ευθυγραμμιστούν, να εξερευνήσουμε το αν υπάρχουν συνέργειε μεταξύ του. Καλωσορίζω λοιπόν την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμείς ως Επιτροπή ΕΚΟΝ είμαστε αποκλειστικά αρμόδιοι για τρεις, τρία κομμάτια της πρότασης, στατιστική, ανταγωνισμός και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Και πιο συγκεκριμένα ο αλφαβητισμός, ο πιστοτικός. Και θα ήθελα από το σχέδιο γνωμοδότησης να τονίσω κάποια στοιχεία. Πρώτα απ' όλα για τα στατιστικά να πω πως η Eurostat δεν θα πρέπει να είναι το θύμα της συγχώνευσης των διαφόρων προγραμμάτων και πιο συγκεκριμένα δίνω κάποιες διευκρινήσεις από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα για να αποδώσουμε μεγαλύτερη σημασία στις σχετικές παραγράφους και προτείνω την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής επιτήρησης με ε, επιχειρησιακές και ε, διοικητικές ε, δαπάνες οι οποίες θα πρέπει ε, να παρακολουθούνται πιο στενά για να ενισχύσουμε και τις αρμοδιότητες της Eurostat. Για την πολιτική ανταγωνισμού, νέες προκλήσεις από, την από τον ψηφιακό κόσμο και εδώ πρέπει να ενισχύσουμε και πάλι την ε, ε, παρακολούθηση της δαπάνης στα πλαίσια του προγράμματος Συνήθειας Αγοράς από το Κοινοβούλιο και για τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υπενθυμίζω πως η χρηματοδότηση για τους μη οργανισμούς που έχουν ασχοληθεί με το θέμα του ε, ε, χρηματοπιστωτικού αλφαβητισμού θα πρέπει να ανοίξει και για νέες αιτήσει από νέες πηγές. Τέλος, στο σχέδιο γνωμοδότησης δεν έχω ακόμα τροποποιήσει το παράρτημα, το έχω κάνει εσκεμένα και στο παράρτημα έχουμε τις επιλέξιμες δράσεις για τη στατιστική. Στο σημείο εδώ δεν έχω καταλήξει, οπότε αν θέλετε να κάνετε προτάσεις θα σας ακούσω με μεγάλη χαρά. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. ΕΛΚ. Η Ρωμανατόντ. Που ήρθα στην ώρα μου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους, ε, τον συνάδελφο κυρίως που παρουσίασε την έκθεση και που προέβαλε τα βασικά στοιχεία. Η κοινή αγορά είναι βέβαια ένα από τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μπορεί να φωλήσει όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι θέλουμε να επιθυμεί να λειτουργεί καλύτερα η κοινή αγορά και να καλύπτει περισσότερους ε, τομείς. Βέβαια υπάρχουν εμπόδια που παρεμποδίζουν την λειτουργία της αγοράς, όπως εμείς θα την επιθυμούσαμε. Και γι' αυτό χαιρετίζουμε την πρόταση Επιτροπής και επιθυμούμε αυτά τα συγκεκριμένα οικονομικά κίνητρα θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Επιθυμώ επίσης η πρωτοβουλία αυτή να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχω πει επανειλημμένα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πιστεύω στον τομέα ε, των στατιστικών. Εκεί μπορούν να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γιατί βεβαίω συγκεντρώνονται τα δεδομένα, αλλά αν δεν τυχάνουν χάνουν σωστή και καλή επεξεργασία, δεν είναι χρήσιμα. Και κάτι άλλο. Όταν μιλάμε για κίνητρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι οι μικρές χώρες ε, δεν ε, θα βρίσκονται σε χειρότερη θέση. Οι μεγάλες χώρες έχουν περισσότερους πόρους και οικονομικούς και σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι μεγαλύτερες χώρες είναι περισσότερο σε θέση να χρησιμοποιούν ε, τα χρήματα για τα ε, προγράμματα. Ε, όπως σας είπα, οι μικρότερες χώρες βρίσκονται σε δυσμενή θέση. Δεν έχουν πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα. Και όσον αφορά στον ανταγωνισμό, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό οι κανένες ανταγωνισμού να την χάνουν αυστηρής εφαρμογής ο αθέμητος ανταγωνισμός εμφανίζεται όλο και περισσότερο σε ορισμένα κράτη-μέλη και μερικές μάλιστα φορές στηρίζεται και από τις κυβερνήσεις αλλά σε τελική ανάλυση οι φορολογούμενοι είναι εκείνοι που επιβαρύνονται με το κόστος αυτών των αθέμητων πρακτικών και μερικές φορές και οι αθέμητες αυτές πρακτικές ε, κατατρώγουν ε, ε, την εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες δεν έχουν ακόμα ακόμα επιβεβαιωθεί και για αυτούς τους λόγους πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την ε, ψηφιακή αγορά. Η δική μας η πολιτική ομάδα θα καταθέσει τροπολογίες και προσβλέπω στην αγαστή συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ ε, για την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, υπερβάσου Μπερές. Θα διαβάσω και πάλι το σημείωμα που Άλφρετσον ετοίμασε για μένα για να τον αντικαταστήσω και σας ζητάει να τον συγχωρέσετε που δεν μπόρεσε να είναι εδώ αυτό το βράδυ. Πιστεύει ότι η γνωμοδότηση που παρουσιάστηκε από τον σαν Σανέδελφο είναι μια μετριοπαθής προσέγγιση πάνω στην οποία μπορούμε να συνεργαστούμε. Θα ήθελε να τον ευχαριστήσει και να τον συγχαρεί θα ήθελε να δώσει μια σύντομη περίληψη σχετικά με το έγγραφο μέλος της ΕΚΟΝ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα γενικά στόχους ε, των, του προγράμματος χρηματοδότησης που πρέπει να ακολουθούν τις βασικές αρχές προστάτευσης του αδύναμου συνδέσμου στην αλυσίδα που είναι συνήθως οι πολίτες ε, και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε ε, να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες για αυτούς. Αυτό θα πρέπει να γίνει και για τις χρηματοδοτικές υπηρεσίες και τους χρήστες ε, που έχουν κακή πληροφόρηση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την προστασία των οικονομικών και νομικών συμφερόντων ε, των χρηστών. Σε σχέση με την ενιαία αγορά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε, να επιτύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Όλες οι πολιτικές γενοσιακές θα πρέπει να προσδιορίζονται από την, ε, τη θεματολόγιο 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη. Πας πάρουμε την ανταγωνιστικότητα σχετικά με τις μικρομεσίες. Οι μικρομεσαίες που εργάζονται παραμύτως χάρη στον τομέα του τουρισμού χρειάζονται πολλές επενδύσεις στον τομέα αυτό για να παραμείνει ανταγωνιστικός συνολικά και ε, σταθερός. Η πρόταση της Κομισιόν μας λέει ότι χρηματοδότηση ε, θα πρέπει να δίδεται όταν υπάρχει υποαξιοποίηση και προτεραιότητα θα πρέπει να είναι ότι η ειδική ενίσχυση δίνεται στις φτωχές περιφέρειες της Ένωσης, αυτές που βρίσκονται ε, στην περιφέρεια, λέει ο κύριος Άλφρεντ Σάντς. Οι φτωχές περιφέρειες ε, είναι, καθυστερούν όταν πρόκειται να ευεργετηθούν από την χρηματοδότηση. Η βελτίωση των στατιστικών είναι σημαντική για την παρακολούθηση της εφαρμογής σε σχέση με τους στόχους, όπως επίσης και το πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ε, χρησιμοποιούνται τα κονδύλια με τρόπο αποτελεσματικό ε, για την ε, διάδοση δεδομένων που να είναι φιλικά προς τους χρήστες, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ε, ε, σχετικά με την ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή οικονομία. Τονίζει ότι ε, βεβαίως δεν είναι η αγορά στόχος, η ευημερία είναι ο στόχος να υπάρχει σε όλες τις περιφερειές, να αυξηθεί η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Ευχαριστώ. Και τώρα για την ομάδα ΟΑΛΔΕ, ο Ραμόν Τρεμόζο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι είναι χαρά για μένα ε, που μπορώ να συγχαρώ τον εισηγητή μας, τον κύριο Λούνες, φίλος όλων και δικός μου. Χαίρομαι που θα συνεργαστούμε για αυτό το θέμα. Ε, συζητάμε το να συστήσουμε ένα πρόγραμμα για την κοινή αγορά, την ανταγωνιστικότητα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα. Συμφωνώ με αυτό που είπαν οι περισσότεροι από εσά ότι το σημαντικότερο επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κοινή αγορά. Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν πολλές αγορές ε, που προσπαθούν να μιμηθούν την κοινή αγορά στην Βόρεια Αμερική, στην Νότια Αμερική, στην Ασία. Ε, εκείνο λοιπόν που μπορούμε να δείξουμε στον κόσμο, αυτό που πραγματικά οι Ευρωπαίοι κατάφεραν καλύτερα από όλα των τελευταίων ήταν η κοινή αγορά, η δημιουργία θέσεων απασχόληση πλούτου και βεβαίω ε, και οι Ευρωπαίοι επέτυχαν ε, το κράτος πρόνοια, ε, το οποίο και αυτό μπορούμε να εξάγουμε στον υπόλοιπο κόσμο. Ω εκ τούτου, οποιοδήποτε πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί για να εμβαθύνει την κοινή αγορά, για μας, για τη δική μας πολιτική ομάδα, είναι προτεραιότητα. Θέλουμε να συνεργαστούμε και με τις άλλες πολιτικές ομάδες για να βελτιώσουμε περαιτέρω την κοινή αγορά. Όταν μιλάμε για στατιστικές, είναι πολύ σημαντικό ε, για όσους χαράσουν πολιτική να έχουν στα χέρια τους ε, τις ε, καλύτερες δυνατές πληροφορίες. Και αν οι στατιστικές, τα στατιστικά δομένα και είναι αρμονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο καλύτερα για τους πολιτικούς, για τους βουλευτές. Άρα δηλαδή και εμείς επιθυμούμε να εκταμιεύονται κονδύλια για να υλοποιηθούν αυτές οι τόσο σημαντικές προτάσεις. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βελτιώσει τα εργαλεία ε, πληροφόρησης, ε, να δρομολογήσει μηχανισμούς όχι μόνο για επιχειρήσεις αλλά και για μεμονωμένα άτομα μαζί με άλλες πολιτικές ομάδες και εμείς ε, θα βοηθήσουμε έτσι ώστε να επιτευχθεί ευρία συνένεση για να βελτιωθεί η κείμενη νομοθεσία. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω να υπάρχει εκπρόσωπος των Πρασίνων ούτε από την ΚΟΕ. Η FTT θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω πως όλα αυτά εμένα μου φαίνονται λόγια του αέρα και πιστεύω ότι καλό είναι οι κυβερνήσεις να μην ανακατεύονται με τις επιχειρήσεις και να μην παρεμβαίνουν. Και αν θέλετε να έχετε ενιαία αγορά, η αγορά οποιοδήποτε τρόπο ρυθμίζει τα δικά τη θέματα η αγορά από μόνη τη. Το καταφέρνει καλύτερα από τι κυβερνήσει, που συνήθω τα κάνουν μουσκεμα όταν προσπαθούν να παρέμβουν στην οικονομική δραστηριότητα. Γιατί δεν καταλαβαίνουν πώ λειτουργούν οι επιχειρήσει. Δεν είναι λοιπόν αναγκαίο κάτι τέτοιο. Α αφήσουμε τι επιχειρήσει να αναλάβουν τα επιχειρηματικά. Αλλά εμεί έτσι κι αλλιώ φεύγουμε και θα το κάνουμε μόνοι μα και μετά θα συγκρίνεται. Όταν εμεί βγάλουμε πολλά λεφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο και όλοι εσεί βρίσκετε σε καθεστώ χρεοκοπία. Um, Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να απαντήσετε στα σχόλια αυτά, όχι απαραίτητα σε όλα τα σχόλια. μπορούμε να έχουμε συζήτηση για τη βιωσιμότητα, θα ήθελα να παραφράσω τον αγαπητό μου ε, φίλο Ραμόν, ζήτω η εσωτερική αγορά, ζήτω η ενία αγορά να την ενισχύσουμε. Και θα λάβω τις ε, τροπολογίες των διαφόρων ομάδων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα προθεσμία 5 Νοεμβρίου για τις τροπολογίες στις 5 το απόγευμα, ε, εξέταση 26-27 Νοέμβρη, 10 Δεκεμβρίου ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ ε, και 21-22 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνεδρίαση σε προχωρημένη ώρα. Θα έχουμε την 5η 25 Οκτωβρίου την επόμενη συνεδρίαση, αυτή την 5η από τις 8 σε 9.45 πάλι μια κοινή με την Econ και την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου από τις 6 ως 7 πέρα της ψηφοφορίας, της συνεδρίασης.